Okay, dear... Ωραία, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Δεν είναι και πολλοί συνάδελφοι παρόντες, αλλά φαντάζομαι σιγά σιγά θα έρθουν. Όπως έλεγα και το πρωί, δεν πρέπει να τιμωρούνται αυτοί που είναι συνεπείς και έρχονται στην ώρα τους. Επομένως, ξεκινήσουμε. Για άλλη μια φορά θα δώσω το λόγο στους διερμηνείς για την ανακοίνωσή τους. Δυστυχώς οι διερμηνείς πρέπει να σας, να σας ενημερώσουν για το γεγονό ότι η διαμάχη με την διοίκηση για τι ε, νέε συνθήκε εργασία, οι οποίε έχουν επιβληθεί μονομερό, συνεχίζεται. Παρά τι διάφορε παραχωρήσει που έχουμε κάνει, η διοίκηση δεν έκανε καμία προσπάθεια για να ε, έρθει σε συζήτηση, σε κάποια συνεννόηση μαζί μα. Δυστυχώ, ε, θα σας ε, ενημερώσουμε ότι θα σταματήσουμε ακριβώς όπως προβλέπετε από το ωράριό μας, δηλαδή στις 6.30 και δεν θα υπάρξει καμία υπέρβαση ωραρίου. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστεί και η Πρόεδρος. Όπως έλεγα και το πρωί, λέει η Πρόεδρος, η διερμηνία είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε, το θεωρούμε πολύ πτυμό. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και πολλά χωρίς εσάς, λέει ελπίζουμε να βρείτε μια λύση η οποία να είναι αποδεκτή και από τα δύο μέρη και η οποία να είναι κατάλληλη. Και μπορώ τουλάχιστον να σας πω ότι σε κάθε περίπτωση εμείς θα έχουμε τελειώσει πριν τις 6.30. Ωραία. Ας περάσουμε λοιπόν στο σημείο το μοναδικό που προβλέπεται στην ημερησία διάταξη για αυτό το απόγευμα είναι η ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Όπως σας είχαμε ενημερώσει και προηγουμένως, έχει δημοσιευτεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο, 30 Μαΐου. Την καλωσορίζουμε ε, καλωσορίζουμε το γεγονό ότι το Creative Europe, η Δημιουργική Ευρώπη, παραμένει ένα πρόγραμμα ξεχωριστό. Αυτό... Το οποίο διατήρησε και το όνομα του, λοιπόν. Και έτσι ταχθήκαμε πολύ υπέρ τη ε, προάσπιση του και στα πλαίσια τη συζήτηση ε, στην Επιτροπή. Αποστήλαμε πολλαπλέ επιστολέ και ξεκαθαρίσαμε ότι δεν επιθυμούμε το πρόγραμμα να χαθεί σε ό,τι αφορά την χρηματοδότησή του σε επιμέρους προγράμματα και ότι πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα λοιπόν αυτό διατηρεί τη σημασία του και γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθησε τις προτάσεις μας και διατήρησε ως αυτό το τέλος πρόγραμμα, το πρόγραμμα Creating Europe. Γίνεται λοιπόν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σήμερα για τις προτάσεις αυτές. Αλλά η Επιτροπή βασικά έχει να μας παρουσιάσει μια μελέτη την οποία εμείς ως Επιτροπή του Κοινοβουλίου δώσαμε εντολή να διεξαχθεί και γι' αυτό έχουμε τον κύριο Λεγκάλ και την κυρία Θεοδόρα Πετούζου. Χαίρομαι που σας καλωσορίζω για να μας παρουσιάσουν τα πιο σημαντικά αποτελέσματα το, της έρευνάς τους. Καλώς επίσης και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μανιέ από το κομμάτι το δημιουργικό και καλλιτεχνικό και από την Γενική Διεύθυνση και τον κύριο στην Γενική Διεύθυνση Connect. Είναι αρμόδιος διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Connect. Ζητώ συγγνώμη. Θα ήθελα καταρχάς να δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονές μας για 10 λεπτά και μετά να ακολουθήσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι έχει να μας πει. Κύριε Λιγκάλα, έχετε το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα και είμαι από την, ε, την ε, σχετική μελέτη που διεξάχθηκε μετά από έντολη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να σα κάνω την παρουσίαση λοιπόν, η οποία είναι αρκετά ξεκάθαρη. Στην παρούσα φάση θα ήθελα απλά να επισημάνω ότι για τους σκοπούς της συζήτησης έχουμε τις συστάσεις ε, πολιτικής και μία γρήγορη ανάλυση διάμεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, της Δημιουργικής Ευρώπης που μπορούμε να συζητήσουμε λοιπόν μετά από την παρουσίαση αυτή. Στόχοι της έρευνας ήταν να παρέχει μια γρηγορη αναλυση ενδιάμεση της ευρωπαικης επιτροπης της δημιουργικης ευρωπης που μπορουμε να συζητησουμε λοιπον μετα απο την παρουσιαση αυτη στοχοι της ερευνας ηταν να παρεχει μια αναλυση τη Δημιουργική Ευρώπη. Εξετάσαμε λοιπόν του στόχου, τη δομή, τη διαδικασία λήψη αποφάσεων και τον αντίκτυπο τη εφαρμογή τη. Το πιο σημαντικό επίση ήταν να δοθούν συστάσει για τα μέλη τη επιτροπή Πολιτισμού για να δημιουργηθεί το μέλλον τη δημιουργική Ευρώπη ω πρόγραμμα. Να σα πω λοιπόν ποια ήταν τα βασικά πορίσματα τη μελέτη μα. Καταρχά η Δημιουργική Ευρώπη έχει θέσει στόχου να καλύψετε τα χάσματα τα οποία υπάρχουν στον ε, κλάδο το δημιουργικό στην Ευρώπη. Καταρχάς υπάρχει απόκληση δημιουργική σε όλη την Ευρώπη σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την ε, ανάπτυξη του πτιακοστικού τομέα στο θέμα του πολιτισμού. Επίσης, ανάπτυξη δυναμικού για τον κλάδο αυτό, ανάπτυξη προσόντων, διεθνή δικτύωση, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και καλύτερη καλύτερα στατιστικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό σε όλη την Ευρώπη. Ένα βασικό πόρισμα επίση είναι ότι ο, συνολικό ε, ε, προπολογισμό για την περίοδο 2014-2015 ήταν ανεπαρκή δεδομένη και τη σημασία του κλάδου στην ε, συνολική οικονομία. 1,46 δις ευρώ για τα 27 κράτη-μέλη για τα 7 χρόνια για να πετύχουμε γεωγραφικά ισορροπημένα αποτελέσματα. Είναι χαμηλός λοιπόν αυτός ο α, προϋπολογισμός δεδομένης της υψηλής, του υψηλού ποσοστού αιτήσεων και χαμηλό ποσοστό επίσης επιτυχίας. Δεν λαμβάνεται υπόψη η διάρθρωση της αγοράς και εδώ βλέπετε σε ένα γράφημα και τα μέσα ενημέρωσης και τον πολιτισμό σε ό,τι αφορά ε, το ποσοστό αιτήσεων 2014-2017. Ένα άλλο σημαντικό σημείο σε ό,τι αφορά τη δημιουργική Ευρώπη. Είναι εξαιρετικό σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη δικτύωσης. Ε, μια ευρωπαϊκή λοιπόν κοινότητα τέτοιων ε, παραγωγών. Και για να γεφυρίσει το χάσμα μεταξύ των πολιτισμικών παραγόντων και των πολιτικών ηθινόντων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δύο σημεία θα ήθελα να τονίσω. Καταρχάς, ε, η, το εργαλείο διευκόλυνσης και εγγύησεων ε, που έχει εγγυηθεί ένα ποσό 50,2 εκατομμυρίων και το οποίο αναμένεται να παρέχει πάνω από 630,4 εκατομμύρια χρηματοδότησης για τις πολιτισμικές μικρομεσαίες. Επίσης, ε, μια άλλη πάρα πολύ σημαντική να σας πούμε ότι δεν υπάρχει επαρκές ανθρωπίνο δυναμικό και περιορισμένο επίσης χρηματικό δυναμικό χρηματοδότηση. Ένα σημαντικό, μια σημαντική πτυχή είναι η λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά τη Δημιουργική Ευρώπη. Η διαδικασία αυτή στην παρούσα φάση κάνει διάκριση μεταξύ δύο μη νομοθετικών πράξεων ε, τη ε, πράξη κατά εξουσιοδότηση και τι εφαρμοστικέ εκτελεστικέ πράξει και αποφασίζεται μαζί με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά πόσο ε, θα υπάρχουν σχετικές πράξεις τέτοιες εκτελεστικές. Φυσικά η διαφορά είναι γνωστή και μπορείτε να διαβάσετε φυσικά λεπτομέρειε στην έρευνά Η βασική διαφορά είναι ότι οι πράξει κατά εξουσιοδότηση απαιτούνται όταν χρειάζονται περαιτέρω νομοθετικέ τροποποιήσει στο βασικό ευρωπαϊκό δίκαιο, ενώ οι εκτελεστικέ πράξει απαιτούνται όταν το ευρωπαϊκό δίκαιο εφαρμόζεται καθεαυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απλά σωστούς και καθολικούς όρους εφαρμογής τη Δημιουργική Ευρώπη χρησιμοποιείται λοιπόν η πράξη κατά εξουσιοδότηση με ένα κατάλογο δικτών ε, που θα πρέπει να τροποποιούνται. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει το πρόγραμμα με τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Κοιτούσαμε λοιπόν το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και διαπιστώσαμε ότι γενικά Υπάρχουν πολιτικέ πτυχέ και ζητήματα τα οποία θα αντιμετωπίζουν στι εφαρμοστικέ πράξει και εκτελεστικέ πράξει και θα έπρεπε να τις τα εξετάζουμε μέσω πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Για παράδειγμα, τροποποίηση του πρόγραμματος εργασίας του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργήσε μια νέα δράση για την ενσωματώση των προσφύγων στο πλαίσιο του μεγάλου κύματος ε, μεταναστών που ξεκίνησε το 2015. Αυτή η εξέλιξη σε πολιτικό επίπεδο προφανώς έχει και πολιτικές επιπτώσεις. που θα έπρεπε να τις κοιτάξουμε σε ιδανικό σενάριο σε πράξη κατά εξουσιοδότηση με τη συμμετοχή του νομοθέτη, του συνομοθέτη. Στο μελλοντικό λοιπόν κανονισμό για τη δημιουργική Ευρώπη θα πρέπει και ο νομοθέτης να αποφασίζει σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή της νομοθεσίας, γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ νομικής βεβαιότητας, συνοχής, δημοκρατικού διαλέγου και διαφάνεια από τη μία, αλλά και ευελεξίας, η οποία χρειάζονται απαραίτητο από την άλλη πλευρά. Θα έρθω τώρα σε ένα άλλο στοιχείο της μελέτης μας που ήταν η συνέργεια μεταξύ της χρήσης του Creative Europe και άλλων ε, προγραμμάτων, ε, όπως το Ορίζοντας 2020, το πρόγραμμα Erasmus. Κάτι σημαντικό εδώ είναι να διαπιστώσουμε ότι οι στόχοι του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη έχουν ενταχθεί σε όλο και περισσότερα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ωστόσο, ε, δεν υπάρχει μια επίσημη στρατηγική ε, για αυτή την αλλαγή, ούτε βέβαια υπάρχει κάποια κοινή προσπάθεια ε, υλοποίηση, δεν υπάρχει κάποια, για παράδειγμα, κοινή στο σελίδα στην οποία να μπορεί να βρει κανεί όλε τι σχετικέ πληροφορίε. Ε, ένα παράδειγμα είναι ότι στον ορίζοντα 2020 έχουμε στόχους σχετικούς με την προώθηση της δημιουργίας των δημιουργών στην Ευρώπη ή επίσης το πρόγραμμα media, το οποίο δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης και εθνικών πόρων. Θα περάσω όμως γρήγορα σε αυτό που νομίζω είναι το πιο σημαντικό για σας σήμερα, που είναι οι προτάσεις μας, οι συστάσεις. Πρώτα απ' όλα, το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να λάβει υπόψη του ε, αλλαγές που έχουν γίνει. Δηλαδή, το γεγονό ότι οι νέοι πλέον καταναλώνουν, αν θέλετε, έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο με διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές αρχές, οι πόλεις, οι περιφέρειες επενδύουν πια στον πολιτισμό ε, και όσον αφορά το ύψος της χρηματοδότησης, αλλά και επίση όσον αφορά τις πολιτικές τους και τις καινοτόμε πρωτοβουλίες τους. Ο ίδιος ο κλάδος της του πολιτισμού ε, έχει και εκείνο αναλάβει κάποιε κοινοτόμε πρωτοβουλίε, ιδίω όσον αφορά τον τρόπο τον οποίο απευθύνεται στην κοινωνία. Και τέλο, το έχουμε πολλέ φορέ συζητήσει, ότι η χρήση των ψηφιακών πλατφορμών έχει αρχίσει να αποκτάει όλο και μεγαλύτερη σημασία και διάδοση και πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας στο μέλλον. Τέλος, δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία επιθυμεί να ενισχύσει την πολιτιστική παραγωγή και να χρησιμοποιήσει τις ε, πολιτιστικές σχέσεις, αλλά και τρίτες χώρες. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε καταλήξει στις εξής συστάσεις. Θα πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός, να γίνει πιο φιλόδοξος. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας πώς θα δημοσιοποιηθεί ε, το πρόγραμμα αυτό και πώς θα δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακος έτσι ώστε να προωθηθούν καινοτόμα προγράμματα έτσι ώστε να ενισχυθεί η διεθνή διάσταση της ευρωπαϊκής πολιτιστική ε, δημιουργία και να αξιοποιήσει η Ευρώπη τον πολιτισμό στις ε, διεθνείς σχέσει. σχέσεις. Προτείνουμε να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο και τέλος να ενισχυθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιείται το πρόγραμμα της Δημιουργικής Ευρώπης για δημιουργικές παρεμβάσεις στην κοινωνία. Κλείνοντα θα έλεγα ότι η πολιτιστική παραγωγή στην Ευρώπη είναι πολύ δυνατή. Υπάρχουν πολλά, πολύ ταλαντούχοι δημιουργοί και πρέπει να δούμε που θα, πώς θα βοηθήσουμε γιατί διαπιστώνουμε ότι μόνο το 0,15% του ευρωπαϊκού προπολογισμού πηγαίνει στον πολιτισμό. Πρέπει να φροντίσουμε αυτό να αυξηθεί στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ συνεκτική η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης σας. Την έχετε όλη στη διάθεσή σας. Διαβάστε την. Περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία. Για το πώς... Ε, θέτουμε προτεραιότητες σε σχέση και με αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να προτείνω να ακολουθήσουμε την διαδικασία όπως σήμερα το πρωί για να ακούσουμε καταρχάς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και στη συνέχεια να κάνετε εσείς ερωτήσεις και προς τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προς ε, εμπειρογνώμονες μας. Να ακούσουμε καταρχά τον κύριο Μανιέ. Μιας και έχει αναλάβει το πιο μικρό τμήμα του προγράμματος. Merci, euh, Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ αξιόματος της Επιτροπής την Επιτροπή Πολιτισμού για την ευκαιρία που μας δίνεται να παρουσιάσουμε την πρόταση της Κομισιόν για το επόμενο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ μαζί με τον Τζουζεμπε Αμπαμόντε για να σας δώσουμε καλά νέα, όπως νομίζουμε. Υπάρχουν τέσσερα βασικά μηνύματα που θέλουμε να περάσουν. Πρώτον, ότι θα υπάρξει συνέχεια. Η Δημιουργική Ευρώπη θα επεκταθεί και θα παραταθεί ως αυτόνομο πρόγραμμα μέχρι το 2027. Δεύτερον, θα υπάρξει ευθυγράμμιση. Η Δημιουργική Ευρώπη θα υποστηρίξει περισσότερο τις πολιτικές προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερως την ενιαία ψηφιακή αγορά και το νέο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο των Πολιτισμών. Τρίτον, καινοτομία. Η Δημιουργική Ευρώπη θα έχει νέες δράσεις για να στρίξουμε καλύτερα τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς και την ευρωπαϊκή δημιουργία. Τέλος, τέταρτο μήνυμα. Επενδύσεις. Η δημιουργική Ευρώπη θα χρηματοδοτείται καλύτερα σε ένα πλαίσιο όπου τα περισσότερα προγράμματα, τα υπόλοιπα προγράμματα κυρίως θα υποστούν περικοπές. Θέλουμε λοιπόν η Επιτροπή πολιτισμού ε, να ικανοποιηθεί, γιατί από την ε, αρχή αυτό που μας έλεγε το λάβαμε υπόψη μας. Λάβαμε υπόψη μας τα αποτελέσματα της ε, διάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος, που έλεγε ότι η Δημιουργική Ευρώπη υλοποίησε τους στόχους, αλλά το πρόγραμμα αυτό υποχρηματοδοτείται. Ε, αυτό επιβεβαιώθηκε από την δημόσια διαβούλευση που έγινε στις αρχές του 2018 και την έκθεση που μόλις πραγματοποιήθηκε για την Επιτροπή Πολιτισμού, τη Δική Επιτροπή. Το πλαίσιο ήταν ευνοϊκό. Ο πολιτισμός ε, αυτή τη στιγμή είναι σε θετική φάση. Ε, ξεκίνησε αυτή η θετική φάση με, το, με την Ευρωπαϊκή Σύνοδο του G7 και του Γκέτεμπορκ, ε, καθώς και τη συνεδρίαση του Νταβός, καθώς ε, και τη συνεδρίαση για την πολιτιστική κληρονομιά το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σα συνεισέφεραν ιδιαίτερω στο να υπάρξει ένα νέο ανανεωμένο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και σα ευχαριστώ γι' αυτό. Η αποστολή του προγράμματο Δημιουργική Ευρώπη θα είναι, όπω και σήμερα, να προωθήσει την ε, πολιτιστική πολυμορφία τη Ευρώπη και την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και δημιουργικού μα κλάδου. Θέλουμε να κρατήσουμε την ε, κοινωνική και εγγενή αξία του πολιτισμού, καθώς και την οικονομική συνεισφορά του. Αυτή η στόχη είναι η ραχοκοκαλιά των δραστηριοτήτων για τον πολιτιστικό τομέα και ισχύει πολύ περισσότερο από ό,τι ποτέ, παρά ποτέ, για την περίοδο 21-27. Μαζί με τον Τζουζέπε σας επαλα... Ε, παρουσιάσω σε τέσσερις φάσεις το πρόγραμμα, την γενική του δομή και τον προπολογισμό του, εν συνεχεία το υποπρόγραμμα πολιτισμό. Ε, συνεχεία το υποπρόγραμμα ΜΜΕ και τέλο το διατομιακό κομμάτι. Για τη δομή και τον προϋπολογισμό είδατε ότι αυτή η δομή είναι περίπου ίδια με την σημερινή. Δύο ε, υποπρογράμματα και ένα διατομιακό. Η βασική αλλαγή είναι το εργαλείο χρηματοδοτικής εγγύησης. Ε, θα περάσει σε ένα επενδυτικό ταμείο με σκοπό να εξασφαλίσουμε ε, στον πολιτισμό τα τραπεζικά δάνεια και αυτό θα είναι ο διάδοχο του σημερινού εργαλείου. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε τρίτε χώρε με βάση τη νέα προσέγγιση ε, στα πλαίσια τη πολιτιστική διπλωματία. Έχουμε βάλει μια γενική ρήτρα σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων που θα διαρθωθεί σε διάφορε δράσει και θα προωθηθεί σε διάφορε δράσει και έχουμε ένα σύστημα παρακολούθηση των επιδόσεων του προγράμματο που θα βασίζεται σε ένα πιο συγκεκριμένο και πιο περιορισμένο αριθμό δικτών, εφαρμόζοντα τη γενική πολιτική που έχουμε για όλα τα προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλο, ο προπολογισμό θα αυξηθεί κατά 27% σε σχέση με την περίοδο 2014-2021. Είδατε ότι θα περάσει σε ένα ε, δισεκατομμύριο 850 εκατομμύρια ευρώ. 1.080.000 για τα ΜΜΕ, 609 για τον πολιτισμό και 160 εκατομμύρια για το διατομιακό κομμάτι. Έρχομαι τώρα στο υποπρόγραμμα πολιτισμός. Εκεί θα θέλαμε να διακρίνουμε τέσσερις κατηγορίες δράσεων. Πρώτη κατηγορία είναι οι δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα. Στο εσωτερικό αυτής κατηγορίας έχουμε τρεις δράσεις που δεν αλλάζουν γιατί λειτουργούν καλά. Ε, εξού και η συνέχεια που θέλουμε να κρατήσουμε. Οι δράσει της συνεργασίας, η υποστήριξη στα δίκτυα και η υποστήριξη στις πλατφόρμες. Προσθέσαμε σε αυτές τις τρεις δράσεις που υπήρχαν ήδη, τρεις νέες δράσεις για την καινοτομία που θέλουμε να επιφέρουμε, η κινητικότητα των καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού που θα δοκιμάσουμε από το 2018 ήδη. Η νέα δεύτερη δράση είναι η εξωτερικοποίηση και των ε, δημιουργικών δράσεων και μια νέα πολιτική για τον πειραματισμό. Αυτές είναι οριζόντιες δράσεις. Πέρα από αυτές τις οριζόντιες δράσεις έχουμε και τομεακές δράσεις που αφορούν συγκεκριμένους τομείς ούτως ώστε να λάβουμε υπόψη μας καλύτερα την ιδιαιτερότητα που έχουν οι αγορές. Ξέρετε μία που είναι η τομεακή, αγορά για την, τομεακή δράση για τη μουσική, το κοινοβούλιο την υποστηρίζει με την παρασκευαστική ε, δράση ε, Music Move. Δεύτερη δράση θα αφορά τα βιβλία με ένα πρόγραμμα μεταφράσεων που θέλουμε να αναθεωρήσουμε και να το κάνουμε πιο αποτελεσματικό. Τρίτον, τρίτη τομεακή δράση θα αφορά την δομή και την ε, πολιτιστική κληρονομιά ε, γύρω από την έννοια του Bau και άλλοι τομείς που θα προσθεθούν καθώς οι ευρωπαϊκές δράσεις θα αναπτύσσονται τρίτη κατηγορία δράσεων, η οποία υπάρχει στο πρόγραμμα πολιτισμό, είναι συγκεκριμένες δράσεις, τι ξέρετε ήδη, είναι οι Ευρωπαϊκέ Πρωτεύουσε Πολιτισμού Φερρυπίν, είναι ο Ευρωπαϊκός ε, τίτλος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ε, τα βραβεία πολιτιστικά βραβεία, οι ε, ευρωπαϊκές ημερίδες ε, πολιτιστικής κληρονομίας που θέλουμε να απτύξουμε και να εξευρωπαίσουμε και να υποστηρίξουμε ε, πολιτιστικούς φορείς Ευρωπαίους όπως η Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Νέων. Αυτά θα υπάρχουν στο υποπρόγραμμα για τον πολιτισμό και τώρα θα δώσω το λόγο στον Τζουζέπε για το υποπρόγραμμα ΜΜΕ. Ευχαριστώ Μισελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τα ΜΜΕ είναι μια πολύ καλή ιστορία επιτυχίας. Θέλουμε να βασιστούμε σε αυτό και όπως είπε και ο Μισελ, από τη στιγμή που υπάρχει το πρόγραμμα, προσπαθούμε να προωθήσουμε την πολιτιστική ποικιλομορφία και την ανταγωνιστικότητα και ιδίω την ανταγωνιστικότητα. Αυτά ισχύουν. Το νέο πρόγραμμα είναι μια μεταξέλιξη του ισχύοντος προγράμματο παρά μια επανάσταση. Το προγράμματα και οι δράσει των προγραμμάτων απαιτούν όμω. ε, εξειδίκευση για να, και αλλαγές για να λάβουν υπόψη κάποιες ε, προκλήσεις όπως το διεθνή ανταγωνισμό που είναι πιο σκληρός παραποτέ. Ο ανταγωνισμός προέρχεται από τα μεγάλα στούντιο, το Hollywood, αλλά προέρχεται και από φορείς που δεν υπήρχαν πριν από λίγα χρόνια, όπως οι παγκόσμιες πλατφόρμες όπως το Netflix ας πούμε. Ε, θέλουμε περισσότερη υποστήριξη για να αυξήσουμε και να ανταγωνιστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα δύο τρία του, του, του, του τρίτα συγγνώμη, του κοινού βλέπουν αμερικάνικες ταινίες και δεν μας αρέσει αυτό. Ποια είναι τα θέματα τα οποία θα στηρίξουμε με το νέο πρόγραμμα. Καταρχάς ε, το κοινό. Μεγαλύτερη εστίαση θα έχουμε στη ζήτηση παρά στην προσφορά. Θα δούμε ποια είναι το, οι ομάδε ανθρώπων που αποτελούν το κοινό. Θα το υποστρίξουμε. Συνεργασία και δικτύωση, δεύτερον, γιατί είμαστε ε, δυνατοί μόνο όταν είμαστε ενωμένοι. Αν είμαστε ενωμένοι θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε ε, με τους μεγάλους παίχτες στην παγκόσμια αγορά. Πρόθεση, διανομή. Τα ευρωπαϊκά έργα θα πρέπει να είναι πιο ορατά και γνωστά για να τα παρακολουθεί ο κόσμο. Γι' αυτό το πρόγραμμα Media ε, θα προωθήσει τα ευρωπαϊκά έργα χάρη και στην οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα. Ε, την ξέρετε πολύ καλά, Πρόεδρε. Το πρόγραμμα Media θα στηρίξει λοιπόν οικονομικά τη διανομή, τις νέες ποσοστώσεις χάρη, που προωθούνται χάρη στην οδηγία για τα οπτακοακουστικά. Και κάτι άλλο, η καινοτομία, το είπε ο Μισελ. Τα, το media ενθαρρύνει την ευρωπαϊκή βιομηχανία να επενδύσει σε νέε τεχνολογίε, όπω ε, εικονική πραγματικότητα, νέε μορφέ, για να προωθήσει την χρήση νέων τεχνολογιών, όπως blockchain, στη διανομή και με σεβασμό των δικαιωμάτων ε, πνευματικής ιδιοκτησίας, το copyright. Το... Θέλω να σας δώσω κάποια προγράμματα τώρα για, το... για το πρόγραμμα Media. Παραδείγματος χάρη το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σινεμά Κινηματογράφων, που ήταν επιτυχές. Ήταν ένα μέσο για να ενισχύσουμε την κυκλοφορία και ορατότητα των ευρωπαϊκών έργων στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κινηματογράφων τα τελευταία δέκα χρόνια βασίστηκε σε ένα πολύ μικρό προϋπολογισμό. Περίπου 10 εκατομμύρια το χρόνο και δεν αλλάζει αυτό από χρόνο σε χρόνο και πιστεύουμε ότι το δίκτυο θα πρέπει να ενισχυθεί ειδικά στις ανατολικές χώρες και σε μικρομεσαίες πόλεις. Η αυξημένη χρηματοδοτική στηρίξη θα επιτρέψει στους κινηματογράφους να κάνουν τις, ε, να επενδύσουν σε καινοτομίες, ε, παραδείγματο χάρη ε, data analytics, για να έχουν καλύτερες πολιτικές πώληση εισιτηρίων, ας πούμε. Επίσης υπάρχουν και άλλα δίκτυα, όπως παραδείγματο χάρη δίκτυα πλατφορμών ε, για video demand που μπορούν να υποφεληθούν από τις οικονομίες κλίμακας, οι κοινοί, ας πούμε, κοινέ βάσεις υποτιτλισμού και δίκτυα ε, φεστιβάλ κινηματογράφων ε, που θα κάνουν και διάφορες εκστρατείες προώθησης ε, και εκτόσεων. Επίσης, η παραγωγή. Θα πρέπει να έχουμε καινοτόμες ιστορίες και είναι σημαντικό επίσης να χρηματοδοτούμε ε, σειρές ε, υψηλού δραματικού περιεχομένου που έχουν μεγάλο κοινό και που μπορούν να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τις αμερικανικές σειρές. Παραδείγματα το Berlin Babylon, γέφυρα, το Σουμπούρα στην Ιταλία, όλες αυτές οι συμπαραγωγές ε, μπορούν να έχουν μεγαλύτερη διεθνή απήχηση και να ταξιδέψουν πολύ πιο εύκολα σε άλλες χώρες. Αν μου επιτρέπεις να δανειστώ λιγάκι την δική σου φρασιολογία, Πρόεδρε, πρέπει να ανταμείβουμε ταινίε οι οποίες μπορεί να έχουν καλύτερη και μεγαλύτερη απήχηση ε, στην, ε, σε διεθνέ επίπεδο. Ε, περιεχόμενο και διανομή. Θα πρέπει να συντονίζουμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Διανομής σε διάφορα εδάφη, να χρηματοδοτήσουμε περισσότερες δραστηριότητε προώθησης και μάρκετινγκ. Είναι πολύ σημαντικό. Μία ταινία που δεν το βλέπει κανένας. Δεν τη βλέπει κανένας. Δεν είναι καλό για τον ανταγωνισμό, ούτε για την πολιτιστική ποικιλομορφία. Τα, οι ταινίε γίνονται για να τις βλέπει ο κόσμος και πέρα από τα σύνορά μας πέρα από τα εθνικά σύνορα και πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης. Κάτι που είναι εξίσου σημαντικό, ότι υπάρχει περισσότερος χώρος για αποτελεσματικότητα. Θα δώσουμε ε, άτοκα δάνεια, επομένως θα μειώσουμε το κόστος του δανεισμού κατά 30% και θα μειώσουμε και το διοικητικό άχθο. διοικητικό ε, κόστος. Παραδείγματο χάρη τα ευρωπαϊκά σινεμά, η ευρωπαϊκή κινηματογράφη Ω φορέας θα παίρνει τα λεφτά και θα διανέμει τα λεφτά σε 2.000 ε, δικαιούχου. Με αυτόν τον τρόπο τα λειτουργικά έξοδα μειώνονται και προωθούνται περισσότερο τα έργα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω και δύο λόγια ε, για, την, για το διατομιακό κομμάτι. Η μεγάλη καινοτομία είναι ε, για πρώτη φορά η συμπερίληψη δράσεων στον τομέα των news media που αφορούν τον πλουραλισμό, την, τη γνώση του πώς λειτουργούν τα ΜΜΕ. Έχουμε εμπνευστεί από τα πιλωτικά προγράμματα της Επιτροπής σας. Είναι πολύ σημαντικό για να συνοδεύσουν τις διαρθωτικές αλλαγές στο νέο κόσμο το ΜΜΕ, ούτω ώστε να δίνουμε νέα ε, που να είναι πολιτιστικά και να μπορεί ο κόσμος να τα βλέπει και με κριτικό πνεύμα, ούτω ώστε ε, να καταπολεμήσουμε και την παραπληροφόρηση. Μια άλλη καινοτομία είναι ένα εργαστήριο ε, για τη δημιουργικότητα που θα Παραδείγματο χάρη γύρι ε, εικονικής πραγματικότητας, ούτως ώστε θα να φέρουμε τον πολιτισμό στα σπίτια των ανθρώπων, ε, ε, σινεμά και αίθουσε θεάτρου θα, θα χρησιμοποιούνται για να οργανώνονται κονσέρτα ε, για να φτάσουμε σε νέο κοινό. Τέλος, ε, το Creative Europe Desk, το οποίο θα χρηματοδοτείται ε, υπό το διατομιακό τομάτι, γιατί είναι η γέφυρα ανάμεσα στην δημιουργική ε, στον δημιουργικό κλάδο και στα προγράμματα. Και θα μας δίνει και χρήσιμη, χρήσιμες απόψεις, χρήσιμα στοιχεία για το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας και τη στήριξής μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τους ε, εμπεριγνώμονες και τον κύριο Μόντα και τον κύριο Μαγιέ και πρωτού ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Να πω την μεγάλη μου χαρά να, προσκα... να ε, καλωσορίσω έξι προσκεκλημένους από την ε, πόλη του Μάντορ, ε, που ήταν και πόλη, η πολιτισμική πρωτεύουσα της Ιταλίας το 2016, αν δεν κάνω λάθος. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην ε, Επιτροπή μας. Ελπίζουμε να παρακολουθήσετε με ενδιαφέρον τις σημερινές μας συζητήσεις. Να επανέλθουμε λοιπόν στην ανταλλαγή απόψεων. Να ξεκινήσουμε τη Σιλβία Κώστα. Έχει το λόγο για πέντε λεπτά, Σερβία. Ευχαριστώ. Άκουσα με μεγάλο, μεγάλη προσοχή τη μελέτη, την εκτιμώ. Γιατί είπατε και θετικά πράγματα ε, και κάνετε και κάποια κριτικά σχόλια, ε, επικριτικά σχόλια. Ε, με ενδιαφέραν και οι τελικές ε, συστάσεις, ε, πολύ ενδιαφέρουσες. Ευχαριστώ τον Μισελ για την παρουσίαση επίσης του προγράμματος. Ε, δεν είμαστε πολλοί. Να ας πούμε ξεκιν... καταρχάς τα θετικά πράγματα. Είναι θετικό το ότι παραμένει αυτόνομο αυτό το πρόγραμμα και έχει τα δύο στοιχεία, τις, τους δύο κλάδους, είναι το διατομιακό κλάδο. Ε, δεν μ' αρέσει αυτό που λέτε όμως για τις, ε, τις αξίες και τη συνοχή δεν είναι σωστή αυτή η τοποθέτηση του Δημιουργική Ευρώπη, νομίζω. Επίσης, είναι προφανής η υποχρηματοδότηση του Δημιουργική Ευρώπη. Ε, είναι σωστή η φιλοδοξία να βάλετε πολλές γραμμές, πολλές τάσεις, αλλά ε, όταν αυτό συνδυαστεί με την υποχρηματοδότηση, αυτό γίνεται αφόρητο τελικά. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Στην πραγματικότητα, κατά απόλυτες τιμές δεν, δεν αυξήθηκε το budget. Ε, αν λάβουμε υπόψη μας και τον προϋπολογισμό, ας πούμε, αυτό το 27% είναι τελώς ανεπαρκές, ας πούμε, συν όλα τα νέα καθήκοντα του Δημιουργική Ευρώπη. Ε, συνολικά είναι πιο ισορροπημένο επίσης ε, το πρόγραμμα και υπάρχει μεγαλύτερη συνάφεια του προγράμματος με την, το, θεμά, το λόγιο για τον πολιτισμό, την ε, οδηγία και τη συνολική προσέγγιση. Ούτω ώστε οι δράσεις να είναι πιο οριζόντιες και να ε, ευθυγραμμίζονται με άλλους κανονισμούς. Αυτό κάθε φορά το λέμε, γιατί αλλιώς όλα είναι κατακαιρματισμένα. Το είπα και χθε στον Επίτροπο Ναύρατσης. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό, ότι δίδεται μεγαλύτερη προσοχή στις αξίες, ε, στο καλλιτεχνικό κομμάτι, μαζί με το οικονομικό κομμάτι και το θέμα του ανταγωνισμού. Ευχαριστώ γι' αυτό. Οι λέξεις έχουν κάποια σημασία. Ε, δεν μιλάτε πια για πρόγραμμα πολιτισμός, ε, αλλά μιλάτε για strand, για κομμάτι. Γιατί αυτή η αλλαγή, θέλω να το καταλάβω αυτό. για τις ε, κατεξιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Θα το συζητήσουμε αυτό. Αλλά μπορούμε να πούμε καταρχήν το εξής. Εσείς εντοπίσατε πολύ σωστά ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες δράσεις για τον πολιτισμό, ας πούμε. Ε, το κομμάτι αυτό το τροποποιείται πολύ περισσότερο σε σχέση με το media. Είχαμε τέσσερις δράσεις, είχαμε τώρα έξι ε, που είναι οριζόντιες, συν τις τομεακές και τις ειδικέ επιπλέον, με τα project και τα σχέδια. Οκ, okay, μπορώ να συμφωνήσω. Γιατί οι οριζόντιε βάζουν κάποια σημαντικά πράγματα, την κινητικότητα των καλλιτεχτών, πάντα το ζητούσαμε αυτό το πράγμα, και μεγαλύτερη διεθνή στήριξη ε, που το συνδέω εγώ με την, διπλωματική, με την πολιτιστική διπλωματία μάλλον. Ε, επίσης ε, κάποια πιλωτικά πράγματα για τη μουσική κτλ. Κάποια, κάποια πράγματα που κάνετε για τη σύνταξη κτλ. Φυσικά όλα αυτά είναι πολύ φιλόδοξα. Όμως, εν τη αυτή περιπτώσει, και για να αποφασίσουμε και εμείς τι θα κάνουμε, στα πλαίσια της συναπόφασης, δεν μπορούμε στο πρόγραμμα να έχουμε στον προϋπολογισμό του ότι θα φτάνουμε μέχρι το τάδε ποσό. Ούτε στον κανονισμό, ούτε πουθενά αλλού μιλάτε για τις ποσοστώσεις. Έτσι. Λέτε το πολύ πολύ, όχι λιγότερο από κτλ. Είναι σημαντικό ο πολιτισμό, α πούμε να έχει υποποσοστώσει ανάμεσα στα οριζόντια, στις οριζόντιες δράσεις και στι τομεακές δράσει. Γιατί έχουμε σχεδόν 12 δράσει σε σχέση με τι 4 που είχαμε. Εάν δεν τα διαιρέσουμε όλα αυτά σωστά, είναι πάρα πολύ δύσκολο οι συνομοθέτε να δώσουμε προτεραιότητα και να πούμε το τάδε είναι πιο σημαντικό από το άλλο. Όλα απαριθμούνται απλώ. Επίση, ένα τεράστιο έλλειμμα, το καταγγείλαμε, και νομίζω και, και η μελέτη το λέει, είναι οι ποιοτικοί δείκτες δεν υπάρχουν. Έχουμε το παρατηρητήριο για τα οπτικοακουστικά, αν και για τα ψηφιακά θα πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα αυτό, και έχουμε και συγκεκριμένες δράσεις. Επίσης, το InvestEU, αυτό ε, είναι οριζόντιο. Πολύ ωραία. Όμως οι πόροι που υπήρχαν στο InvestEU μπήκαν στο γενικό προϋπολογισμό. Έτσι, καλό είναι αυτό. Όμως, σε ένα κανονισμό καλό θα ήταν να πούμε πώ η Κομισιόν βοηθάει για το πώς ας πούμε, θα χρησιμοποιήσουν οι δικαιούχοι ας πούμε, αυτά τα ποσά του InvestEU. Γιατί αλλιώς τα πράγματα είναι ξεκάρφωτα έτσι. Για το media ε, χαίρομαι για τις καινοτομίε, ε, τα δίκτυα, ε, τα φεστιβάλ. Αλλά δεν υπάρχει καμία αναφορά στα οπτικοακουστικά στο ψηφιακό, συγγνώμη. Ε, στις, παλιά μιλούσαμε για ταινίε ε, μεγάλου μήκους, μικρού μήκους, όλα αυτά εξαφανίστηκαν. Επίσης, ε, δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στα μεγάλα σχέδια και τα μικρά σχέδια. Κακό αυτό για μας. Ε, διατομιακά και κλείνω. Εστιάνομαι σε οριζόντιες δράσεις, παλιά δεν ήταν έτσι. Και τελευταίο ερώτημα. Το θέμα της διακυβέρνησης. Ε, μάθαμε ότι ότι αν δεν υπάρχει μία διακυβέρνηση όπως κάναμε για το ευρωπαϊκό έτος, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε μία διακυβέρνηση με τους stakeholders και την αρμόδια ε, γενική διεύθυνση. Ούτως ώστε να υπάρχει μία ολοκλήρωση πόρων και προγραμμάτων και σχεδίων. Έχουμε του άλλου κόντσμο, τον ορίζοντα, το κοινωνικό α, ταμείο. Δεν υπάρχει μια διασύνδεση ανάμεσα σε αυτά τα προγράμματα. Όλα αυτά είναι καταγερματισμένα. Ποιο θα ήθελε λοιπόν τώρα να απαντήσει. Έχετε παρατηρήσει να κάνετε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία ping-pong για να είναι λίγο πιο ζωντανή η συζήτηση. Wer möchte von Ihnen? Λοιπόν, για το ερώτημα που μου θέτεται για το γεγονό ότι δεν μιλούμε πλέον για υποπρογράμματα αλλά για strands. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι απλώ μια νομοτεχνική αλλαγή. Μα είπαν ότι είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον όρο. Χωρίς να αλλάζει τίποτα στην ουσία. Όσον αφορά τώρα την, για, την κατανομή του προϋπολογισμού στα διάφορα strands. Αυτό φαντάζομαι θα γίνει μέσω των κατευθυντηρίων γραμμών και του ετήσιου προγράμματος εργασίας. Και αυτό χρειάζεται έτσι ώστε να μην έχουμε ε, μια άκαμπτη δομή, να μπορούμε να ε, προσαρμόζουμε τις διάφορες δράσεις. Είναι κάτι το οποίο ήδη κάνουμε. Όσον αφορά τους δείκτες. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να αναθεωρούμε τους δείκτες που χρησιμοποιούμε στο τρέχον πρόγραμμα και το αποτέλεσμα αυτής της αναθεώρησης θα το χρησιμοποιήσουμε στην επόμενη περίοδο. Όσον αφορά τώρα το επενδύοντα στην Ευρώπη, InvestEU, πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία για τον τομέα του πολιτισμού να το αξιοποιήσει για να βρει επιπλέον χρηματοδότηση. Ιδιαίτερα, μάλιστα, εάν το εγκαιοδοτικό σύστημα, το ε, συνεχίσει να λειτουργεί με την ταχύτητα που λειτουργεί. Στο πρόγραμμα επενδύοντας στην Ευρώπη αναφέρεται ρητά ο τομέας του πολιτισμού και μάλιστα εάν λάβουμε υπόψη μας, κάνουμε τον υπολογισμό, ότι και, και λάβουμε υπόψη μα ότι το πρόγραμμα τη εγγύηση δανείων είναι ξεχωριστό, θα δούμε ότι η αύξηση είναι 34%. Μια σημαντική αύξηση. Βεβαίω είναι μια δυνητική αύξηση, δεν είναι κάτι το οποίο ε, έχει συμβεί ακόμα, αλλά μπορεί να γίνει. Όσον αφορά τα προγράμματα συνεργασίας, πράγματι δεν υφίσταται στη νέα νομική βάση αυτή η διάκριση μεγάλου και μικρού project, αλλά εμείς θα τη διατηρήσουμε. Ε, βεβαίως τα μεγάλα προγράμματα συνεργασίας δημιουργούν μια γενικότερη δομή στον κλάδο, ενώ τα πιο μικρά προγράμματα συνεργασίας μπορούν να βοηθήσουν μικρότερους δημιουργούς. Ε, θα γνωρίζετε ότι και με τι τωρινέ ε, κατευθυντήριες γραμμές μας και με την τωρινή μας προσέγγιση προσπαθούμε να κρατάμε μια ισορροπία ανάμεσα στα μεγάλα και τα μικρά project και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Για το θέμα που θίξατε για το media και το πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα τώρα που δεν έχουμε πλέον τα λεγόμενα υποστηρικτικά μέτρα, schemes. Μετά την αξιολόγηση που κάναμε, είδαμε ότι αυτή η δομή του προγράμματος ήταν παροχημένη. Ότι τελικά με αυτό το σύστημα με τα σκιμ οδηγούμασταν σε μια λειτουργία του προγράμματος όπου το ένα σκιμ ήταν τελείως αποκομμένο από το άλλο. Επομένως τώρα προσπαθούμε να έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία. Ε, ε, δεν θα ήταν εφικτό να έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των παραγωγών και των διανομέων κτλ. εάν κρατούσαμε τα ΣΚΙΜ. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν για μεγαλύτερη ευελιξία και για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις εξελισσόμενες ανάγκες του κλάδου, αποφασίσαμε να καταγράψουμε ε, κάποιες βασικές προτεραιότητες και να έχουμε αντίστοιχες δράσεις για όλες τις προτεραιότητες αυτές, οι οποίες δράσει όμως θα εστιάζονται σε όλη την ε, αλυσίδα από την παραγωγή μέχρι τη διανομή του πολιτιστικού αγαθού. Κάτι αντίστοιχο προσπαθούμε να κάνουμε και με τους δείκτες. Τώρα στο media, στο νέο media, προσπαθούμε να έχουμε λιγότερους δείκτες, οι οποίοι να, έχουν, να είναι πιο συναφείς με τα είδο των δράσεων που χρηματοδοτούμε πια μέσω του προγράμματος media και επίσης να είναι εφικτό να τους μετρήσει κανείς με βάση τα δεδομένα που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Τι σημαίνει αυτό. Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να καλύπτουν όλη την αλυσίδα από την παραγωγή μέχρι τη διανομή ε, και την προώθηση και όλα τα στάδια αυτά. Ένας τέτοιος δείκτης είναι ε, η αξιολόγηση που θα κάνουμε κατά πόσο ένα πρόγραμμα τελικά βοήθησε ε, να αυξηθούν οι δεξιότητες στο, σε έναν επαγγελματικό τομέα. Αντί για παράδειγμα να μετρούμε ε, μηχανιστικά απλώς τον αριθμό των δικαιούχων. Γιατί πράγματι οι συμπαραγωγές είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να ενισχύσουμε τη διασυνοριακή συνεργασία στον πολιτισμό. Θέλουμε να αυξήσουμε επίση ο αριθμό των ε, προσώπων που ε, είναι οι αποδέκτες αυτών των πολιτιστικών αγαθών. Αυτό επίσης θα μπορέσουμε να το μετρούμε. Και τέλος, θα πρέπει να αξιολογούμε με τους δείκτες μας πόσο αυξάνεται η ε, δημοσιοποίηση και η γνώση για τα ευρωπαϊκά πολιτιστικά αγαθά. Ευχαριστώ κύριε Βέντα. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ήδη... Ο κύριο δεν θα επαναλάβουμε αυτά που είπε συνάδελφο η κυρία Σιλβία Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρουσίασή σα και συμφωνώ απόλυτα. Να αναφέρω μόνο ένα άλλο στοιχείο. Καταρχά, ε, θα πρέπει να είναι φιλόδοξο ο προπολογισμό για την δημιουργική Ευρώπη. Και έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούμε να πετύχουμε χωρίς ιεράρχηση των στόχων και θα πρέπει λοιπόν να μπει αυτό και στην πολιτική υποστήριξη της ε, Δημιουργικής Ευρώπης. Ένα σημαντικό στοιχείο της ε, μετάβασης ε, της, της του κλάδου είναι ο οπτή οπτικοακουστικός για όλους αυτούς που συμμετέχουν στην, στον κλάδο. Και θα πρέπει η Ευρώπη να δείξει ηγεσία στον τομέα αυτό για να αφαλίσει όλες τις υπηρεσίες του κλάδου. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι ο κλάδος. 4,4% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και 4 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Αλλά σε σχέση με άλλους κλάδους φαίνεται ότι είναι υποτιμημένο στη χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τις συστάσεις λοιπόν της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έκθεση Έλερ και Μοργάνο, θα πρέπει να υπάρχει σωστή χρηματοδότηση για την δημιουργική Ευρώπη και να κοιτάξουμε να στραφούμε προς την οριζόντια ενσωμάτωση του προγράμματος σε άλλα προγράμματα όπως και ο ορίζοντας 2020 παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο για τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών για το πρόγραμμα 2021-2027, θα πρέπει να τεθούν στόχοι και κατευθυντήριες γραμμές ε, και η γραμμή δράση θα πρέπει να είναι σαφής για να υπάρχει μια σχετική σταθερότητα για όλα τα μέρη που συμμετέχουν στον κλάδο αυτό και όπως γνωρίζετε σε ό,τι αφορά τη μουσική. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τομεακή προσέγγιση και για τον τομέα αυτό μετά από την προσέγγιση του 2020. Εγώ υποστηρίζω αυτό το κίνημα Music Moves Europe εξ αρχής ε, για την ενίσχυση της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά ειδικά τη μουσική. Σε ό,τι αφορά όμως τη χρηματοδότηση, ο τομέας της μουσικής δεν ωφελήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό από το 2014 και μετά από τη Δημιουργική Ευρώπη. Μόνο 3%. 0,15% του συνολικού προσυμπολογισμού της Ένωσης έχει αφαιρεθεί σε project μουσικής. Με το νέο που το θα κληθούμε να βρούμε λύσεις για αποτελεσμό, για παράδειγμα, στο Art Europe, προκειμένου τελικά να επεκταθούν τα προγράμματα αυτά και για άλλα για άλλες γλώσσες. Εδώ λοιπόν να κύπτουν ε, ερωτήματα. Ποια λύση μπορούμε να βρούμε σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της διαδικασίας υποτιτλισμού. Σας ευχαριστώ κύριε Βεντάλη, πρόεδρος. Κύριε Μόντα, κύριε Μανιέ. Γιατί, τις υποτιτλισμό. Δεν ε, αποκλείουμε τη δυνατότητα να βρούμε χρηματοδότηση για τον υποτιτλισμό. Το 2019, για παράδειγμα, αν επιτρέπει ο προπολογισμό, θα υπάρξουν νέε δράσει υποτιτλισμού πολιτισμικού περιεχομένου. Με άμεση επιδότηση προς το άρτε, προς το κανάλι. γιατί το ΆΡΤ παρέχει συνοριακή πολιτισμική σύμβολη χωρίς ε, καμία σύγκριση με κανένα άλλο πρόγραμμα και φυσικά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης. Κύριε Μανιέ, για τον υποτιτλισμό να προσθέσω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα τεθεί άμεσα ενδεχομένω και για το θέατρο και για διάφορες άλλες τέτοιες τέχνες ε, ε, παραστάσεις. Ε. Είναι ένα θέμα το οποίο ήδη το αναμένουμε για το ερώτημα για τη μουσική τώρα. Να ευχαριστήσουμε καταρχάς το Κοινοβούλιο για την υποστήριξη που μας έδειξε σε ό,τι αφορά το Music Moves Europe. Να αξιοποιήσουμε τα τρία χρόνια που μας χωρίζουν από την ε, προθεσμία εφαρμογής του προγράμματος για να κάνουμε κάποιο πειραματισμό. Κύριε Βέντα, νομίζω ότι στο τρέχον πρόγραμμα να σας πω ότι δεν είμαστε στο 3%. 15-20% της δημιουργικής Ευρώπης χορηγείται προς το κλάδο της μουσικής. Δεν είναι 3%. Πρόκειται λοιπόν για μια υποστήριξη η οποία όμως δεν είναι τόσο διαρθρωμένη, είναι πιο πολύ μια ενίσχυση κατά περίπτωση σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα αυτό, το Music Moves Europe. Η μουσική κινεί την Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ η Ελκά. Ευχαριστώ Πατρά. Να ξεκινήσω με τα συνολικά θέματα περί χρηματοδότηση. Γιατί αυτό επηρεάζει φυσικά τη δημιουργική Ευρώπη. Νομίζω ότι ήταν καλή η πολιτική προθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να αυξηθεί η χρηματοδότηση. Ιδιαίτερα μετά από αυτά ακούσαμε από την Συνολομέλεια για μείωση του προπολογισμού μετά τον Brexit και το καθεξής. Ήταν ανοησίες. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γεγονός ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή, ως Επιτροπή Πολιτισμού θα θέλαμε πιο πολλά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσευξάνει την πρόταση του Οτινγκέρ και αυτό είναι σημαντικό για όλα τα δημιουργικά κινήματα. Προφανώς ε, είναι Καλό να υπάρχουν πιο πολλοί πόροι, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε μια απόπειρα τουλάχιστον να υπάρξει μια κίνηση. Να περάσω στο όλο θέμα το οποίο θέσαμε και προηγουμένω ψηφιακή επανάσταση και τι σημαίνει για τον πολιτισμό. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο το Netflix και όλοι πάλι φορεί φορείς στην ψηφιακή αγορά που παρουσιάζουν τεράστιες προκλήσεις. Εξακολουθούμε να έχουμε πολλές ε, πειρατικές ιστοσελίδες που κάνουν streaming και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Χρειαζόμαστε επίσης πιο πολλά μοντέλα για να γράφεται κανείς σε ιστοσελίδες. Μέχρι να το πετύχουμε αυτό δεν θα υπάρχει πρόοδος. Πιστεύω ότι όταν ε, κοιτάμε την μελέτη, αυτό που βλέπουμε ότι 7,5% ε, των Ευρωπαίων εργαζομένων ε, εργάζεται στον δημιουργικό τομέα και επίσης ότι εδώ υπάρχει απασχόληση νεολαίας ιδιαίτερως. Πιο πολύ από κάθε άλλο κλάδο, ιδιαίτερα στη μουσική αλλά και σε άλλους δημιουργικούς κλάδους. Οι νέοι είναι αυτοί που είναι ένθερμοι και θέλουν να εργαστούν εκεί. Είναι σημαντικό λοιπόν και στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τμήμα αυτό της οικονομίας μας και του πολιτισμικού τοπίου. Να περάσουμε τώρα στο Music Moves Europe Φέτος είχα την ευκαιρία να παραβρεθώ στις Κάνες για να τονώσω και τη σημασία της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Αυτό είναι θετικό. Και με κάλεσαν να παρουσιάσω ένα καινούργιο έργο στις Κάνες. Ήταν πραγματικά θαυμάσια εμπειρία. Έχει κανείς ε, μία διεθνή αίσθηση πολλών νέων από όλες τις υπήρους ε, πολύ παγκοσμίο το κλίμα και ενθουσιώδεις νέοι άνθρωποι δεν είναι τόσο, αν θέλετε, πνευματικό ζήτημα. Είναι πιο πολύ συναισθηματική αντίδραση, ξέρετε, γιατί πάντα μιλάμε για τις τιμές στην Ευρώπη, για τις κρίσεις που ταλανίζουν την Ευρώπη, τι μέσα στην Γερμανία, Brexit, αλλά το να υπάρχει κάπου και μια καλή αίσθηση είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τους νέους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε κι εσείς κάποιο σχόλιο να κάνετε. Κύριε Μανιέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Τρούπελ για την υποστήριξή της και το Music Move of Europe που είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια. Ε, χαιρόμαστε που αυτή, αυτός ο ενθουσιασμός, αυτή η φιλοδοξία είναι κοινή. Μάλιστα, για να δω από εδώ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Οι περισσότερες ερωτήσεις αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα-δύο πράγματα. Ε, ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας σε τι συνεισέφεραν. Όπως είπατε, είναι πολύ σημαντικό για την απασχόληση των νέων. Αλλά σκεφτείτε που διενεργείται. Ε, στις πόλεις μας. Ε, δεν μπορούμε να εκχωρήσουμε και να αναθέσουμε σε εξωτερικούς φορείς εκτός Ευρώπης ε, το κομμάτι αυτό. Και με αυτόν τον τρόπο ε, εμπλουτίζει τις πόλεις μας και τις κάνει πιο ελκυστικές και δημιουργεί ε, ένα θετικό κλίμα. Συνεισφέρει λοιπόν ποικιλόμορφα. Το αναφέρουμε και στη μελέτη, αλλά και σε άλλες μελέτες αναφέρεται. Έχει και ευρύτερη επίπτωση όμως. Και πολύ σωστό αυτό που είπατε για το θέμα το συγκεκριμένο στη δική σας παρέμβαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να περάσουμε στα υπόλοιπα μέλη. Σκιώδης άλλους δεν βλέπω. Η Κριστίνα Λιμπάτσκα έχει τώρα το λόγο για δύο λεπτά. Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχουμε αρκετή χρηματοδότηση για όλα αυτά τα προγράμματα. Όχι μόνο για τη Δημιουργική Ευρώπη, αλλά και για το Εράσμου, για τον Ορίζοντα και για πολλά άλλα προγράμματα. Δεν αρκεί η χρηματοδότηση. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που έχει σημασία είναι οι συνέργειε των προγραμμάτων, ούτω ώστε να έχουμε μεγαλύτερη, ε, τη μεγαλύτερη δυνατή επίπτωση με του περιορισμένου πόρου. Θα ήθελα λοιπόν να δημιουργηθούν συνέργειε ανάμεσα στη Δημιουργική Ευρώπη, τον Ορίζοντα και, τον, ε, και το έρασμό. Κάποιο από εσά είπε ότι τα δύο τρίτα των θεατών και ακροατών μας παρακολουθούν αμερικανικές ταινίες και σειρές. Και αυτό δεν είναι καλό. Όχι απλώς δεν είναι καλό, είναι καταστροφικό. Γιατί όχι μόνο είναι κακό για το δημιουργικό τομέα, το δημιουργικό κλάδο, αλλά είναι πολύ κακό και για την οτροπία, ειδικά των νέων. Γι' αυτό ακριβώς αυτές οι συνέργειες ανάμεσα στην κινητικότητα των παιδιών και των νέων στο πρόγραμμα Εράσμους και την κινητικότητα των ανθρώπων που εργάζονται στον πολιτιστικό τομέα. Φερρυπίν είναι πολύ σημαντικό. Ένα παράδειγμα από την Αυστρία. Τα κέντρα τα εκπαιδευτικά και τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης ε, συστεγάζονται στο, στους ίδιους χώρους με πολιτιστικούς φορείς κτλ. Ε, αυτό κάνει στην Αυστρία. Καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε ο κύριε Μόντε. Ε, Ευχαριστώ για αυτό το σημείο. Για μας αυτό ήταν μεγάλη πρόκληση, οι συνέργειες, η συνέργεια ανάμεσα στα προγράμματα. Είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος αυτός για να πετύχουμε περισσότερο, περισσότερα πράγματα με προπολογισμού περιορισμένους, παρότι έχουμε κάποιες αυξήσεις εδώ και εκεί. Έχουμε μια εμπειρία ενθαρρυντική στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έτους. Συνειδητοποίησαμε ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα είναι σαφές και ότι θα πρέπει να συμμετέχουν διάφοροι συμμετέχοντες. Είναι πολύ εύκολο να υπάρξει κινητοποίηση των μέσων. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα στα πλαίσια ενό ετήσιου προγράμματο όπω το Ευρωπαϊκό Έτο ε, Πολιτιστική Κληρονομιά, αλλά αυτό μπορεί να γίνει πιο μακροπρόθεσμα στα πλαίσια τη διαχείριση όλων των προγραμμάτων. Γι' αυτό ακριβώς στα, περισσότερε βάσει νομικές βάσεις βάλαμε κάποιες διασταυρούμενες παραπομπές και αναφορές ε, ενώ ε, προς άλλα προγράμματα. Σε κάθε πρόγραμμα δηλαδή γίνονται παραπομπές σε άλλα προγράμματα. Ακριβώς αυτό είναι σημαντικό. Η νομική βάση να είναι ξεκάθαρη, ούτως ώστε να ενημερώνονται οι πιθανοί αποδέκτες το συντομότερο δυνατό για να ξέρουν τι παίζει. Voilà, αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Δεν ξέρω αν όλοι θα διαβάσουμε τόσο ενθουσιασμό τις νομικές βάσεις μας, αλλά αν το κάνουν οι πιθανοί εταίροι, θα δουν ότι κάθε φορά προσπαθούμε να βάλουμε και στόχους που μπορούν να υλοποιηθούν και από άλλα μέσα. Παραδείγματο χάρη, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτου Κληρονομιά, συνειδητοποίησαμε ότι η διάσταση η επιστημονική του πολιτισμού, τη πολιτιστική κληρονομιά, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό θα υπάρχει επίση στο επόμενο ε, και στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Επίση, οι συνάδελφοι τη Γενική Διεύθυνση που ασχολούνται με τι εξωτερικέ δράσει ε, συνειδητοποίησαν ότι τα πολιτιστικά προγράμματα είναι επωφελή στου στόχου του. Και στις, ε, ναι, στην νέα νομική βάση των εξωτερικών προγραμμάτων θα υπάρχει αναφορά στον πολιτισμό. Αποτέλεσμα, αν θέλουμε να έχουμε συνέργειες, έχουμε την νομική βάση για να το κάνουμε. Ενώ προς το παρόν ε, οι σημερινές νομικές βάσεις δεν μας διευκολύνουν, μας δυσκολεύουν. Αυτό μας απασχόλησε πάρα πολύ, ε, εγγύψαμε πραγματικά σοβαρά επί του θέματος αυτού και θα το δείτε σε όλες τις νομικές βάσεις αυτό το στοιχείο. Σας ευχαριστώ σε ό,τι αφορά την αλληλεπικάλυψη προγραμμάτων από διάφορα προγράμματα μάλλον και σε ό,τι αφορά την ωφέλεια διαφόρων προγραμμάτων στο ίδιο έργο όπου καλείται κανείς να εξετάσει ποιο πρόγραμμα τεράστι ταιριάζει καλύτερα. Αυτό αν είναι άρα για το Creative Europe, αν είναι κάποιο άλλο πρόγραμμα, εδώ θα πρέπει να θα πρέπει να πούμε ότι θα έχει νόημα να μην είναι αυτός ο οποίος θέλει να κάνει την αίτηση που θα πρέπει να βγάλει άκρη από την πληθώρα προγραμμάτων, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το κρατός μέλος θα μπορούσε να διαπιστώσει κάθε φορά αν ισχύει για παράδειγμα ορίζοντας 2020. και να μην χρειάζεται να κατατίθενται διαφορετικές αιτήσει για διάφορα προγράμματα. Γιατί, σε πάση περιπτώσει, απευθυνόμαστε και στον ε, απλό πολίτη. Αν θέλουμε λοιπόν να υπάρχει εγκάρσιος χαρακτήρα των προγραμμάτων, θα πρέπει ο κόσμος που κάνει τέτοια αιτήματα να μην χρειάζεται να τα βγάζει πέρα από το λαβύρινθο των προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη από εθνικέ υπηρεσίε. Και σε περίπτωση αμφιβολία να ζητείτε η βοήθεια και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί για τον ορίζοντα 2020 δεν υπάρχει εθνική υπηρεσία αρμόδια. Θα πρέπει και από διοργανωτική άποψη να υπάρχει σωστή οργάνωση. Η κυρία Σόιτροβα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις παρουσιάσεις. Έχω μια παρατήρηση και μια ερώτηση. Ξέρετε ότι εμείς ποτέ δεν μας είμαστε ικανοποιημένοι με το ύψος του προϋπολογισμού. Το ερώτημα όμως πάντα είναι πώς μπορούμε να το χρησιμοποιούμε ε, αποτελεσματικά. Το ερώτημα. Με την έκθεσή σας αναφερθήκατε και είπατε ότι χρειάζεται περισσότερο δημοκρατική συζήτηση. Είπατε, εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερο δημοκρατικό έλεγχο Όσον αφορά το, πολι... το έτος πολι... ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, ε, πρέπει να πω ότι είναι επιτυχημένο το πρόγραμμα μεν, όμως αυτό που δεν είναι ικανοποιητικό είναι η χρηματοδότηση. Χρειάστηκε να χρηματοδοτήσει 29 έργα, όμως σε αυτά τα 29 έργα δεν υπήρχε γεωγραφική ισορροπία μόνο ένα ε, έργο ερχόταν από την κεντρική Ευρώπη, ήταν στην Ουγγαρία προκειμένου. Τώρα όσον αφορά το πρόγραμμα Media, με την βοήθεια της ανάπτυξης διεξιοτήτων. Εννοούμε επίσης και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ε, στον κινηματογράφο. Κατά την άποψή μου χρειάζεται να δώσουμε εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα, να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα βραβεία, τα ευρωπαϊκά βραβεία, το βραβείο Λούξ για παράδειγμα. Είναι πιστεύω μια ευκαιρία που δεν την αξιοποιούμε όσο πρέπει, ούτε επίσης την εκπαίδευση στον κινηματογράφο. Μήπως θα μπορούσατε να μου δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το τι σκοπεύουμε να κάνουμε στο μέλλον με αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ξεκινώ από αριστερά. Κύριε Λεγκάλ, ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ναι, εν συντομία. Για τη δημιουργική συζήτηση, για την ε, δημοκρατική συζήτηση και το δημοκρατικό έλεγχο. Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στις πράξεις κατά εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις. Ε, εδώ, για να το συνοψίσουμε. Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι η Δημιουργική Ευρώπη είχε εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και μάλιστα με θετικό τρόπο. Το πρόγραμμα, για παράδειγμα, για την ενσωμάτωση των ε, μεταναστών. Ήταν ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Θα ήθελα λοιπόν να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία να επιδεξίσουμε ε, ευελιξία και αυτό διατηρείται πραγματικά ως δυνατότητα ακόμα και σε δύσκολες πολιτικές ε, συνθήκες και συγκυρίες. Ε. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός προκειμένου η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να εργαστούν προς την επιτεύξη των νέων αυτών στόχων και να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει και κοινό πολιτικό βάρος, αν θέλετε, γιατί είδαμε με την πρωτοβουλία Music Moves Europe ότι πρόκειται για ένα κοινό εγχείρημα, μια κοινή πρωτοβουλία, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προκαθορίσει προπαρασκευαστικές δράσεις ε, και γι' αυτό λοιπόν προτείναμε να μπουν όλα αυτά στις ε, πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Επιτρέποντας παράλληλα τη δυνατότητα για πιο πολύ δημοκρατικό έλεγχο. Αυτή θα ήταν η θέση μας ε, εν συντομία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε την πρόταση αυτή και Εμεί ε, θέλουμε πιο πολλές ε, πράξεις κατεξουσιοδότηση και λιγότερε εκτελεστικέ πράξει. Ε, κύριε Μανιέ, για την πολιτιστική κληρονομιά και ο κύριο Μπαμόντα για τα μίντια. Sur la question, για το ερώτημα που μου θέσατε για τα προγράμματα συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτου. Πράγματι, μόνο ένα από τα 29 έργα είχε ως ηγετικό εταίρο μια χώρα της κεντρικής Ευρώπης. Θα διαπιστώσετε όμως ότι σε πολλά άλλα προγράμματα, σε πολλά άλλα project υπήρχαν εταίροι ε, που, που προέρχονται από την κεντρική Ευρώπη. Θα παραδεχτώ ότι υπήρξε ε, ένα έλλειμμα γεωγραφικής ισορροπίας, αλλά αυτό ήταν εντονότερο όσον αφορά τις ηγητικούς εταίρους σε σχέση με το αν δούμε το πρόγραμμα συνολικά. Θα γνωρίζετε ότι την προκήρυξη εκτελέσεως ενδιαφέροντος χρειάστηκε να την ολοκληρώσουμε πάρα πολύ γρήγορα γιατί είχε υπάρξει μια καθυστέρηση στο πρόγραμμα εξαιτία της νομοθετικής διαδικασίας, επομένως δεν υπήρχε αρκετός χρόνος προετοιμασίας, επομένως ήταν λογικό ότι οι καλύτερες προτάσεις να έρθουν από χώρες που είχαν μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτά. Έχετε δίκιο, δεν είμαστε ικανοποιημένοι και εμείς, όμως του λεχθέντος πρέπει να σας πω, ότι η ποιότητα των project που εγκρίθηκαν ήταν εξαιρετική και ήδη είδαμε τα αποτελέσματα. Αυτό είχα να απαντήσω σε σχέση με το Ευρωπαϊκό της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ και για την ερώτηση, γιατί μου δίνει την δυνατότητα να σας δώσω ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί να υπάρξει καλύτερο συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων. Πράγματι με το νέο πρόγραμμα Media θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την εκπαίδευση. Με το νέο πρόγραμμα μας τον Οκτώβριο θα κάνουμε μια προκήρυξη με την οποία θα ζητούμε να υπάρξει μια καταλογογράφηση των ευρωπαϊκών κινηματογραφικών έργων που είναι μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και θα μπορούσαν να διατίθενται στα σχολεία. Εμείς λοιπόν θα υποστηρίξουμε την δημιουργία του καταλόγου και ο Μισελ θα μας δώσει ε, το κατάλογο του με τους εκπαιδευτικούς και θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε αυτό το δίκτυο εκπαιδευτικών ε, για τη διανομή. Πάντως, για να απαντήσω άμεσα στο ερώτημά σας και συνοπτικά, ναι, βεβαίω θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την εκπαίδευση των κινηματογράφων. <clears throat> Eh, Ευχαριστώ. Αν προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε το τι ακούσαμε και στην εισαγωγή, στην παρουσίαση της ε, μελέτης και στην ε, συζήτηση που ακολούθησε, ε, το συμπέρασμα νούμερο ένα που προκύπτει είναι ότι ο πολιτισμός θα πρέπει να χρηματοδοθεί καλύτερα. Ταυτολογία είναι αυτό, αυτονόητο είναι, το λέμε, αλλά το μήνυμα δεν περνάει. Καινοτομίε, πλατφόρμες, πρόσβαση σε περιεχόμενο, μεγαλύτερη ορατότητα, διεθνής διάσταση. Έτσι, τίτλοι είναι αυτοί που πετάω και θα μπορούσα να παραθέσω πάρα πολλού άλλου. Όλα αυτά, χωρί έναν τρόπο για να τα υλοποιήσουμε, κίνδυνο, ο κίνδυνος είναι στο εγγύς μέλλον να γίνει αυτό που φοβάστε, ότι κάποια προγράμματα θα έχουν αύξηση εις βάρος κάποιων άλλων προγραμμάτων. Επομένω, θα παραμείνουμε σε αδιέξοδο και μπλοκαρισμένοι. Γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί με απασχολούν τρία προβλήματα. Καταρχά, μέτρηση των επιπτώσεων. Πώ γίνεται αυτή η μέτρηση, μέσω δικτών. Τώρα, κάποιοι δείκτε είναι ξεκάθαροι, ενώ άλλοι δείκτε, επιτρέψτε μου να σα πω, για τον πολιτισμό, ε, που συνδέονται με πούμε τον αριθμό των θεατών. Είναι νομίζω πολύ περιοριστική. Γιατί γιατί αν εγώ δεν κάνω άλλες επενδύσεις για να ξεπεράσω κάποια όρια, όπως είπε η συνάδελφος προηγουμένως, τότε θα μείνω σε αυτά που έχω σήμερα. Και δεν θα δώσω καθόλου κίνητρα για να αυξηθεί ο αριθμός, ας πούμε, των θεατών ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, για να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα πολιτιστικά και τη δημιουργικότητα. Επίσης, συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε την νομική βάση, αλίμονο, αλλά μαζί με την νομική βάση χρειάζεται και ένα εργαλείο, ούτω ώστε να γίνει εφαρμοστέα η νομική πράξη, γιατί ακόμα και αυτή η νομική βάση θα παραμείνει γράμμα και ενώ περιεχομένου. Συγχωρήστε μου την έκφραση. Ευχαριστώ πολύ. Και περνάμε τώρα στην ε, τελευταία, ε, στο τελευταίο γύρο. Κύριε Μανιέ, κύριε τα είπατε όλα. όλα τα σχόλια των ομιλητών για το ότι δεν ε, με εκπλήσουν καθόλου. Είναι μουσική στα αυτιά μου, γιατί εγώ αυτό πιστεύω. Μπορεί να θεωρείτε ότι η αύξηση στον προπολογισμό είναι περιορισμένη, αλλά πετύχουμε λοιπόν παραπάνω αφού αυτό θεωρείτε Ναι, βεβαίω, λέει η πρόεδρο, να το προσπαθήσουμε. Ναι, να σας πω και κάτι άλλο για τα εργαλεία. Τι προβλέπετε συγκεκριμένα μετά την νομική βάση, ούτω ώστε να υπάρξει αυτή η σύνδεση ανάμεσα στα προγράμματα. Γιατί αλλιώς μόνο με το να υπάρχουν διασταυρούμενες παραπομπές μέσω των νομικών βάσεων δεν αρκεί να συνδεθούν, ε, να υπάρξει σύνδεση με τα άλλα προγράμματα. Καταλάβατε πολύ καλά τι εννοώ. Είναι γνωστή η Επιτροπή μας για τα ανοιχτά λόγια που χρησιμοποιούμε. Ποιο θέλετε να απαντήσει, να απαντήσει στο ερώτημα αυτό, κύριε Μανιά, κύριε Μόντα. Κοιτάξτε, ναι. η νομική βάση είναι, αν θέλετε, η βασική σύμβαση που έχουμε. Είναι αυτό που μας επιτρέπει να κάνουμε δαπάνες από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, που θέτει τα, τους όρους. Είναι ένα, μια, ένα νομικό εργαλείο όμω. δεν είναι ένα εργαλείο για την επιχειρησιακή διάρθρωση του προγράμματο. Από εκεί και πέρα έχουμε τα επιχειρησιακά εργαλεία. Είναι οι κατευθυντήριε οδηγίε για την κάθε μια από τι δράσει, τι οποίε πράγματι πρέπει να απλοποιήσουμε γιατί είναι και αυτό ένα ζητούμενο, και οι οποίε κατευθυντήριε οδηγίε περιγράφουν πώ εφαρμόζονται, πω υλοποιούνται οι διάφορε δράσει και μετά για να υπάρχει η απαραίτητη ευελιξία και στην υλοποίηση του προγράμματος, να μπορεί το πρόγραμμα να ε, προσαρμόζεται στις αλλαγές, έχουμε τα ετήσια προγράμματα δράσης. Και στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης κάθε χρονιάς βλέπει κανείς ποιες προκηρύξεις θα γίνουν ε, και όλα, όλα τα υπόλοιπα. Αυτό το σύστημα έχει και πλεονεκτήματα και, και μειονεκτήματα. Το μειονέκτημα του είναι ότι κάπως φορτωμένο, δηλαδή ότι κάθε χρονιά πρέπει να ετοιμάζουμε όλα αυτά τα έγγραφα, τα οποία είναι ένα φόρτο εργασία που θα προτιμούσαμε να μπορούσαμε να μειώσουμε. Έχει όμω και το πλεονέκτημα ότι εξασφαλίζει τη χρηστή διοίκηση, την ορθή διαχείριση των πόρων. Κάτι το οποίο είναι μια, ένα απόλυτο ζητούμενο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζετε ότι υπάρχει το ελεγκτικό συνέδριο, ότι δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να ε, πληγεί το κύρος αυτών των προγραμμάτων εξαιτίας περιπτώσεων απάτης ή άλλων τέτοιων περιστατικών. Το ερώτημα λοιπόν που, είναι, που τίθεται είναι πώς μπορούμε να βρούμε μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ το, της χρηστής διοίκησης του προγράμματος και των ε, απαιτήσεων που θέτουμε στους δικαιούχους. Γιατί πράγματι αυτή τη στιγμή είναι κάπως βαρύ το πρόγραμμα, ε, δημιουργεί ένα συγκεκριμένο φόρτο. Όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούμε την απέτηση για νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών. Ορίστε η απάντησή μου λοιπόν. Η νέα νομική βάση είναι πιο απλή και ε, λιγότερο μακροσκελής από την προηγούμενη. Είναι αυτό μια γενικότερη επιδίωξη που έχουμε ακολουθήσει στην Επιτροπή. Όλα τα νέα προγράμματα να είναι ε, πιο σύντομα, πιο συνοπτικά έτσι ώστε οι νομικέ βάσεις πραγματικά να στέκονται στι ουσιαστικέ προτεραιότητε και από εκεί και πέρα να έχουμε άλλα έγγραφα τα οποία να εξειδικεύουν τι προτεραιότητε αυτέ. Ε, το ακολουθήσαμε στο δικό μα πρόγραμμα, αλλά το ίδιο κάνει η Επιτροπή για όλα τα προγράμματά τη. Τώρα ίσω μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε αυτό, γιατί δεν είμαι σίγουρο ότι μπορώ να το καταλάβω. Έχουμε ήδη κάποια εργαλεία τα οποία δουλεύουν, έχουμε τι επιδοτήσει, οι οποίε αποδίδονται μετά από μια προκήρυξη. Ο κύριο Αμπαμόντα μιλάει καταρχά και μετά θα πάρει τη στο λόγο, Σίλβια. Ωραία. Από ό,τι φαίνεται δεν κατάλαβα ποια ήταν η ερώτησή σας λοιπόν. Και αν δεν καταλάβω την ερώτηση, δεν θα σα δώσω απάντηση ικανοποιητική. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μήπω μπορείτε να αναδιατυπώσετε την ερώτησή σα τότε. Τώρα να πάρει το λόγο η Σίλβια για να διευκρινίσει. Προσπαθήσω. Μπέρδεψα τα μικρόφωνα. Δεν σας διακόπτω. Θέλω να σας εξηγήσω γιατί καταλάβα ότι δεν ε, εννοήσατε τι λέγαμε και δεν λάβαμε σωστή απάντηση. Δεν αρκεί να μας πείτε ότι με βάση τη νομική βάση θα έχουμε αυτούς τους, αυτές τις συνέργειες. Κάτι που προκύπτει και από εμά αλλά και από τη μελέτη είναι ότι πολλοί από αυτούς τους επιπλέον πόρους ε, δεν αρκούν, ειδικά για τον πολιτισμό. Ε, διαπιστώσαμε ότι πηγαίνουν και σε άλλα προγράμματα, ειδικά στο Ευρωπαϊκό Έτος ε, Πολιτισμού. Δεν αρκούν αυτές οι παραπομπές. Πρέπει να έχετε κάτι περισσότερο, περισσότερο στις νομικές βάσεις, να μιλήσετε με άλλες γενικές διευθύνσεις και να βάλετε διασταυρούμενες παραπομπές στους άλλους κανονισμούς. Για να μην γίνονται αυτές οι συνέργειες μόνο ad hoc, έτσι. Γιατί αλλιώ, έχουμε 12 δράσει. Εάν θέλετε να κρατήσουμε και τι 12 δράσει, εφόσον δεν έχουμε αρκετά λεφτά, θα πρέπει να μα πείτε ποια δράση έχει η προτεραιότητα. Δεν μπορείτε να μα λέτε έχουμε τι συγκεκριμένε τι οριζόντιε και τι τομεακέ. Να κάνετε κάποια κλάστερ, α πούμε, δράσεων. Ε, για τον πολιτισμό, Φερρυπίν. Ε, Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν, γιατί έχουμε τι 12 δράσει, δεν υπάρχει καμία ιεράρχικη προτεραιότητα στι δράσει αυτέ και λείπουν και δείκτε. Τι γίνεται λοιπόν, χάο. Σας ευχαριστώ και νομίζω ότι στο σημείο αυτό ενδεχομένως να χρειαστεί και περαιτέρω συζήτηση. Ενδεχομένως ε, να πρέπει να υπάρχει και προσαρμογή ή διευκρίνηση στις ε, τροπολογίες. Ελπίζοντας να μας ακολουθήσει και το Συμβούλιο, θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω και τους δύο μας ε, εμπειρογνώμονες για την πολύ καλή και ωφέλιμη παρουσίαση και νομίζω ότι καταλάβατε από τις παρεμβάσεις μας ότι όχι μόνο διαβάσαμε την ε, έρευνα σας αλλά και θα την αξιοποιήσουμε στο μέλλον. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παμόντα και τον κύριο Μανιέ για το γεγονός ότι ήταν εδώ σήμερα Θα παραμείνουμε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνία μαζί σα, προκειμένου να βελτιώσουμε περαιτέρω τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι μόνο θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι κυρίως θέμα των κρατών μελών, γιατί αυτό εξαρτάται, από αυτά εξαρτάται το πόσο βαθιά θα βάλουν ο χέρι στην τσέπη. Θα δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε τελική ανάλυση και χαίρομαι και προσβλέπω στη μελλοντική συνεργασία και εύχομαι κυρίως στον εισηγητή και στους κοιόδης ε, να πάνε όλα καλά σε ό,τι αφορά την ε, έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και το μοναδικό λοιπόν που έχω ακόμα να σας ανακοινώσω, μιας και δεν έχω τίποτα άλλο στα διάφορα, είναι ότι η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει η χώρα 11 Ιουνίου μεταξύ 9 μέχρι 12.30 και το απόγευμα από 3 μέχρι 6.30. Το απόγευμα στις 11 Ιουλίου να σας πω ότι θα διοργανωθεί και η ακρόαση για την πολιτισμική ατζέντα και θα χαιρόμουν ε, ιδιαίτερος να δω πιο πολλούς ε, εδώ συναδέλφους από ότι σήμερα. Αυτό λοιπόν θα μπορούσατε να μεταφέρετε ως μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευγενικά πρώτος, σε ευχαριστεί και τους διερμηνείς που ολοκλήρωσαν και δύο ώρες νωρίτερα και ελπίζουμε να μην έχουν και περαιτέρω δουλειά σήμερα. Σας εύχομαι λοιπόν καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ.